συντάξεις. Θέμα που υποσχολεί όλους μας φαντάζομαι. Κυρία Εισηγήτρια έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Κρούζ, χαίρομαι που είστε εδώ παρούσα. Θα ήθελα να ξεκινήσω να προβαίνονται σε ένα άλλο σχόλιο. Άκουσα την Άντα Ντίγμαντς που είναι στην ορδική ε, καμπίνα διερμηνεύσει, η οποία θα μας εγκαταλείψει έχει, και θα βγει στη σύνταξη, έχει χαρακτηριστική φωνή και θα μας λείψει. Και χαίρομαι που την άκουσα απόψε να διερμηνεύει. Ελπίζω αυτά που είπα να μην αφαιρούνται από το χρόνο αγόρευσής μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής της εκθέσεως θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους τον συνάδελφό μου, τον κύριο Τόμας Μαν, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη συνεργασία που είχαμε, που ήταν και ευχάριστη και καρποφόρα. Θέλουμε όλοι να έχουμε μια βιώσιμη σύνταξη, επαρκή, αυτό θέλουμε όλοι. Όμως ε, οι συντάξεις είναι ευθύνη των κρατών μελών και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη ως Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα σαν Ευρωκοινοβούλιο. Η συντάξεις αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πρόγραμμα σταθερότητας και εθνικών μεταρρυθμίσεων. Και αυτό που μετράει για μένα και για τους συναδέλφους είναι η κοινωνική συνιστόσα των συντάξεων. Πώς θα φροντίσουμε ούτω ώστε στα άλλα κράτη-μέλη οι συντάξεις να μπορούν να διατηρηθούν σε καλό επίπεδο. Τώρα έχουμε μία πυραμίδα πληθυσμιακοί, αντεστραμμένη. Υπέρχουν περισσότεροι ηλικιωμένοι με καλή ηλικία και λίγα άτομα που χρηματοδοτούν ε, τη σύνταξη. Υπάρχει γύρανση του πληθυσμού. Ένα τρίτο του πληθυσμού είναι πάνω από 55. Ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης είναι πάνω από 55 ετών. Στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά συστήματα συνταξιοδοτικά Έχουμε συστήματα του πρώτου πυλώνα που εκφράζουν την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι πολύ σημαντικό στο μέλλον. Αλλά με γυράσκοντα πληθυσμό αυτό σημαίνει μεγαλύτερες πιέσεις επί των νέων, μεγαλύτερες πιέσεις επί της αλληλεγγύης. Η αύξηση των δαπανών του προπολογισμού ε, είναι κάτι που επηρεάζει το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά και βλέπουμε ότι στις χώρες που υπάρχει έλλειψη χρημάτων και υπάρχει μεγάλο χρέος δημόσιο, ότι εκεί οι πρώτες μειώσεις, οι πρώτες περικοπές που γίνονται ακριβώς αφορούν τις συντάξεις. Αυτό πρέπει να αποφευθεί. Όχι μόνο πρέπει κανείς να εργάζεται περισσότερο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και περισσότεροι άνθρωποι που εργάζονται για να λυθεί το πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη αυτοί που δεν εργάζονται σήμερα, που είναι άνεργοι. Θα πρέπει περισσότεροι άνθρωποι προχωρημένης ηλικία να εργάζονται, θα πρέπει να υπάρχει και ευέλικτη δυνατότητα εργασία και να υπάρχει και σωστή προσαρμογή, ούτω ώστε να μπορεί ο κόσμος να συνεχίζει να εργάζεται. Από αυτή την έποψη ο πρώτος πυλώνας είναι σημαντικότατος. Για τις χώρες όμως που εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα, εκεί Έχουμε συνταξιοδοτικούς φορείς όπου οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες συνεργάζονται. Αλλά και εκεί ασκούνται πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω της κακής κατάστασης της αγοράς των μετοχών και των ομολόγων και εκεί βέβαια ισχύει και το πρόβλημα προκύπτει από τη γύρανση του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ε, θέλει τώρα να ασχοληθεί με το επίπεδο των κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών ταμείων. Αυτή δεν είναι σωστή απάντηση. Δεν είναι η ορθή λύση, δεν αρκεί αυτή η λύση, διότι στις χώρες όπου δεν υπάρχουν καλά ομόλογα ε, και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις συντάξεις. Κυρία Κρούζ, εσείς θα πρέπει να μας δώσετε προσανατολισμούς, προτάσεις. Κλείνοντας, Τρίτος πυλώνας, και κλείνω εδώ, ασφάλειες. Νομίζω ότι χρειάζονται να γίνουν περισσότερα εκεί. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε τι έχουμε ήδη και τι οικονομίες έχουμε κάνει σε αυτόν τον τομέα. Μετά, τελευταίο σημείο, η κινητικότητα. Η ελεύθερη κυκλοφορία ε, δεν μπορεί να επιτρέπεται παρά μόνο αν δεν υπάρχουν, δεν δημιουργούνται προβλήματα. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ρία για την εξαιρετική έκθεσή σου για ε, όλα αυτά που είπες ιδιαίτερα για, το, ε, αυτά που είπες στο τέλος και για το τις ασφάλειες και την υποχρέωση για το Solvency 2. Είναι ε, δύσκολο να φανταστούμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και στις συντάξεις. Κάνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσέξτε γιατί ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά στις, στα διάφορα κράτη-μέλη. Μην τα μπερδεύετε με την ασφάλιση ζωής. Χρειάζονται πάρα πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων χωρών. Ε, το κόστος όφελος είναι διαφορετικά, διαφορετικό στο κάθε ε, κράτος μέλος. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε και να λέμε solvency δύο για όλους τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε η συγγήτρια, οι συντάξει κατά κύριο λόγο με τις ιδιαιτερότητές τους είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Βεβαίως το θέμα αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο γιατί βιώνουμε μια εποχή κρίσης και μας απασχολεί όλους γιατί τον πρώτο πυλώνα πραγματικά θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, να μην δίνονται μοναχά ελάχιστες ε, συντάξεις. Το δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας είναι διαφορετικός με τα ερωτηματικά του και εκείνο που είναι σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορούμε ε, εκτός από τους ε, ηλικιωμένους να, φρο... να, πείσουμε και τους νέους να αποταμιεύουν τρόπον την είναι πολύ δύσκολο ε, να κάνουμε κάτι τέτοιο και βεβαίως ε, η έκθεση δεν είναι σοσιαλιστική όπως θα τη θέλαμε εμείς αλλά είναι ένας καλός συμβιβασμός και συμφωνώ μαζί της. Ο κύριο ε, Πάσκα, όπω είπα και πριν, ε, δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε κάποιον που έχει ξαναμιλήσει σε προηγούμενη συζήτηση. Ευχαριστώ. Οι σταθερές ε, βιώσιμε συντάξει, αποτελούν εχέγγυο για όσους είναι σε παραγωγική ηλικία, ότι μπορούν δηλαδή να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη για όταν σταματήσουν να εργάζονται τα αναδυναμητικά συστήματα δεν έχουν λειτουργήσει. Και βέβαια το επόμενο πρόβλημα είναι η ύφεση και η χρεοκοπία των τραπεζών. Άρα τα συγκεκριτικά προγράμματα δεύτερου πυλώνα ε, που στηρίζονται σε προϊόντα της χρηματοψηφιακής αγοράς θα πρέπει να ελέγχονται καλύτερα για να μην ε, κινδυνεύουν, να μην ε, είναι ακάλυπτοι σε κινδύνους οι συνταξιούχοι. Θα πρέπει λοιπόν να παρέχονται σωστές πληροφορίες και για το ποσό που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό και για το κίνδυνο, τα ρίσκα τα οποία μπορεί να αναλάβει ο συνταξιούχος και θα πρέπει να αποφασίσει για το ποια ε, ρίσκα θα ε, λάβει για τη μελλοντική του σύνταξη ή όχι. Eh, η Καρτίκα Λιωτάρ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ρία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τις καταστροφικές προτάσεις Κομισιόν σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα ε, τη συντάξεων επιχειρήσεων. Πολύ ξεκάθαρα λέτε ότι η Κομισιόν πρέπει να σεβαστεί τα συστήματα των κρατών μελών. Για τον πρώτο πυλώνα γιατί δεν έχουμε την ίδια ε, σαφήνεια. Εμείς πρέπει να απορρίψουμε πάση θυσία την πρόταση από την Ολλανδία για να ε, σχετίζεται δηλαδή σύνταξη με τα έτη εργασίας να αποτρέπεται η πρόορη συνταξιοδότηση. Όλα αυτά είναι κακές προτάσεις, ε, αλλά δεν είναι καν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα αποφασίζει αυτά τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να αγκιόνται οι συντάξει είναι ένα ε, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Λέει όμως η Κομισιόν ότι χρειάζεται δεύτερος και τρίτος πυλώνας για αξιοπρεπείς συντάξεις. Με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σέβεται το άρθρο 114 της συνθήκης όπου λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραβιάσει, να θίξει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Λυπούμε γιατί για τον πρώτο πυλώνα δεν λες ε, ξεκάθαρα ρία ότι δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος ευχαριστώ κύριος Μπέκερ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή που αναφέρει στο μέλλον των συντάξεων στην Ευρώπη. Βεβαίως είναι θέμα προτεραιότητας και βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το πρώτο πυλώνα και από εκεί και πέρα συμπληρωματικός να είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ξέρουμε ότι αυτές ήταν διεξιδήσεις ε, διεκδικηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες δεν ε, ε, ολοκληρώθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν τελικά. Έχουμε όμως ένα κοινωνικό μοντέλο στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με τις, το θέμα των συντάξεων. πολλοί μιλάνε και για τη φτώχεια σχετικά. Όχι, η φτώχεια και ο κοινωνικός από είναι άλλο θέμα κοινωνικής πολιτικής. Όμως εδώ για τις συντάξεις σίγουρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε πέρα από λαϊκισμούς. Το οφείλουμε στην επόμενη γενιά να κάνουμε κάτι τι. Η κυρία Ζούπερ 33 ετών σκέφτεται το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή η έκθεση που εκφράζει κοινοβουλευτικέ ιδέε οδηγούν σε δύο βασικού στόχου. Να προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, στη μεταρρύθμιση των συντάξεων και να εξετάσουμε και τις ε, διάφορες επικουρικές ιδιωτικές συντάξεις στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα. Δεν θέλουμε να αυξήσουμε ε, την ηλικία συνταξιοδότηση, Θέλουμε όμως να μπορεί ο κόσμος να γυράσκει με γήτροπο. Και δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα εκείνων που έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα από δεκαετίες δουλειά. Θέλουμε τα ρύθμιση σωστή και να έχουν σωστή σύνταξη και άνεση και να μπορούν να χαλαρώσουν οι συνταξιούχοι. Θα πρέπει να είναι βιώσιμες οι συντάξεις. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τις εισφορές των εργοδοτών και να κινηθούμε σε δημόσιο σύστημα, θέλουμε να εξασφαλίσουμε και ότι και οι τράπεζε θα συμβάλλουν. Διότι μόνο κέρδη βγάζουν από τι ιδιωτικέ συντάξει τράπεζε. Θέλουμε μια καθολική προσέγγιση στον φάτ συντάξει, που θα βασίζονται αυτέ οι συντάξει στην αλληλεγγύη. Δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τον κόσμο να αγοράσει ιδιωτικέ συντάξει. Είναι προβλήματα δημογραφικά αλλά και κατανομή του πλούτου και δικαιοσύνη. Στην Πορτογαλία η Τρόικα είναι υπέρ των, των εργάζονται οι άνθρωποι μέχρι την ηλικία των 67. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και θα είναι κρίσιμη σημασία η μάχη που θα δώσουν οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η ε, κυρία Κρού, Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ε, πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μενράιτεν και τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική συνεργασία τους και διότι ενέκριναν το βασικό πνεύμα της Λευκής Βίβλου. Όταν παρουσιάσαμε τη Λευκή Βίβλο το Φεβρουάριο του 2012, θέλαμε να δείξουμε το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε με βάση το ιστορικό και το πλαίσιο που ανέφερε η κυρία Όμεν του γυράσκοντος πληθυσμού και των οικονομικών περιορισμών να δείξουμε λέγω ότι τα συνταξιδοτικά μας ταμεία παραμένουν και βιώσιμα και ικανά να χορηγήσουν ε, αξιοπρεπή σύνταξη στους συνταξιούχους. Η Λευκή Βίβλος περιγράφει το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε το χρόνο που ξοδεύεται στην εργασία με τη συνταξιοδότηση και να γίνονται και περισσότερες οικονομίες στα επικουρικά ταμεία. Προτείνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα βάσει παλαιών διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη και με τους ενδιαφερομένους φορείς. Και όλα αυτά συνέβαλαν ε, στη συζήτηση που έγινε το 2012 για την, δια, αλληλεγγύη μεταξύ γενεών και την ε, υγιή γύρανση του πληθυσμού. Πρέπει να αξιολογήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του προσδόκιμου ζωής και έτσι να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους και οικονομική ανεξαρτησία στους ηλικιωμένους. Καλωσορίζω και τη συμφωνία του Κοινοβουλίου που πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξουν επικουρικά ε, συνταξιωτικά ταμεία και να σχεδιαστούν του το τρόπος, ούτως ώστε να μην εμποδίζουν την κινητικότητα στην αγορά εργασία. Εξεφράστησαν κάποιε ανησυχίε στην έκθεση όσον αφορά τη διαφύλαξη τη συμφωνία ε, των δημοσίων συντάξεων του πρώτου πυλώνα. Σα διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει, όσο περιεγράφει και στην έκθεση επαρκείας περί συντάξεων του 2012, ότι η δημόσια συντάξη του πρώτου πυλώνα θα πρέπει και θα παραμείνουν βασική πηγή των εισοδημάτων των ηλικιωμένων στο προβλεπόμενο μέλλον. Και από όταν δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο η Λευκής Βίβλο έχουμε πετύχει καλή πρόοδο όσον αφορά αυτή την εφαρμογή κυρίως ε, αυτά που αναφέρονται στην Λευκή Βίβλο ε, συμπεριλαμβάνονται και στάσεις των διαφόρων χωρών. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τους άντρες και τις γυναίκες να εργάζονται περισσότερο. Το πνεύμα της εκθέσεως της κυρίας Όμεν Ράιτον επίσης επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από τα συνταξιωτικά μας ταμεία και να γίνουν τα σωστά βήματα για τη διαφύλαξη του μέλλοντός τους. Όμως, για να πετύχουμε το διτό στόχο επάρκειας και βιωσιμότητας, που είναι φιλόδοξη στόχη, χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες από όλους κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εμπλεκομένους φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε πάρα πολύ, ευχαριστώ συνάδελφοι. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Ρία Όμεν Ρόιτεν, έξοχη και σημαντική έκθεσή τη. Καλύτερε ευχέ όχι μόνο προ την Ολλανδική καμπίνα, προ όλου του διερμηνεί. Του εύχομαι κάποια μέρα μια πολύ καλή συνταξιοδότηση και χαρούμενη συνταξιοδότηση. Έκθεση του κυρίου Γκάιερ για περιφερειακή στρατηγική για βιομηχανικές περιοχές Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θέμα. Γιέν Γκάιερ, έχετε το λόγο.